Έχουν ζητήσει το λόγο πρώτη η κυρία Μορβάη. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι έλλειψη σεβασμού να αρχίσω να μιλάω κάτω από αυτές τις συνθήκες. Δεν είναι σεβασμός και των ε, <clears throat> εκλογέων μας. Παρακαλώ δώστε τρία λεπτά στους αποχωρούντες να αποχωρήσουν και να ξεκινήσουμε μετά από αυτό. Δεν θέλω να μιλήσω σε τέτοιες συνθήκες. Εντάξει, αλλά παρακαλώ και τους συναδέλφους να αποχωρήσουν από την αίθουσα σεβόμενοι και τους αγορητές. Αν θέλετε να περιμένουμε ένα-δυο λεπτά, πρωτού ξεκινήσουμε με τις επεξηγήσεις ψήφων. Eh. Να ξεκινήσουμε. Επεξηγήσει ψήφων για τη Συμφωνία Σταθεροποίηση και Σύνδεση Ευρωπαϊκή Ένωση Κωσυφοπεδίου, σύσταση τη κυρία Λούνατσεκ. Η κυρία Μορβάη έχει το λόγο για ένα λεπτό. Παρακαλώ. Ε, ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. η Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης με το Κωσφοπέδιο ε, θα την είχαν υπερψηφίσει. Α, διότι η διεθνής κοινότητα έχει καταφέρει να εξασφαλίσει την πλήρη αυτονομία για την σερβική μειονότητα στο Κωσφοπέδιο Και το συμπέρασμα το οποίο μπορώ εγώ να αντλήσω είναι ότι οι Ούγγροι που ζουν στη Σερβία θα έπρεπε και αυτοί να έχουν το δικαίωμα της πλήρους αυτοδιάθεσης. Τελικά όμως δεν μπόρεσα να ψηφίσω ναι, γιατί <clears throat> προσωπικά έχω διαπιστώσει ότι οι πρόσφυγες από το Κόσοβο έρχονται στην Ουγγαρία και διαμαρτύρονται για το πλήρες χάος και την πλήρη διαφθορά που ισχύει εκεί. Θα ήταν θαύμα λοιπόν αν οι συνθήκες οι οποίες υπήρχαν τότε έχουν αλλάξει μέχρι τώρα και είναι τόσο διαφορετικές όπως περιγράφει αυτή η έκθεση. Ευχαριστώ. Χωρίς μικρόφωνο. Δεν για ένα λεπτό παρακαλώ. Δεν είναι παρόν. Δεν είναι παρόν. Ντέβα. Α, εδώ είναι. Κύριε, δεν θέλετε να λάβετε τον λόγο. Θέλω, λέει ο κύριος Δέβα. Κύριε Πρόεδρε, το θέμα της σταθεροποίησης του κοσφοπεδίου είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για τις ε, ρυθμίσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια και σταθερότητα στα Βαλκάνια και στη Μεσόγειο. Το Κωσυφοπέδο έχει περάσει μεγάλη αναταραχή και είναι παράδειγμα χώρας η οποία πέρασε από μια μεγάλη αντιπαράθεση σε κατάσταση ειρήνευσης. Έχουμε ξεχάσει, έχουμε παραγνωρίσει κάποια από τα θέματα που έχουν να κάνουν με το κοσφοπέδιο εδώ και πολύ καιρό γιατί μας απασχολήσαν άλλα θέματα σε άλλες περιοχές. Αλλά αυτό είναι θετικό. Μην ξεχνάτε <clears throat> ότι ξαναφέραμε το θέμα μιας χώρας που έχει υποφέρει πάρα πολύ και πάλι στο προσκήνιο και θα πρέπει να εκτείνουμε χείρα φιλίας προς το κοσφοπέδιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ υπεστήριξα την, την πρόταση ψηφίσματο. Βέβαια δεν είναι όλα θετικά στο κοσφοπέδιο. Υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία μπορούν να τύχουν επίκριση, υπάρχουν πολιτικά προβλήματα, περιπτώσει ε, <clears throat> διαφθοράς, μη πλήρους επιβολής του κράτου δικαίου στο κοσφοπέδιο. Από την άλλη πλευρά, εμεί θα πρέπει να συνεργαστούμε με το κοσφοπέδιο, θα πρέπει να εργαστούμε για να μπορέσει να γίνει πλήρω μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και εμείς θα πρέπει να ασχοληθούμε με τις ε, γειτονικές χώρες εκεί. Αν δεν υπάρχει καμία ελπίδα για τους πολίτες αυτών των χωρών, αν δεν υπάρχει ελπίδα για οικονομική σταθεροποίηση και πολιτική ε, ασφάλεια, τότε είναι υποχρεωμένοι να φύγουν από τη χώρα τους και να προσπαθήσουν να έρθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να ξεφύγουν από αυτές τις αντιπαραθέσεις. Γι' αυτό είναι προς το συμφέρον μας να εξασφαλίσουμε τη σταθεροποίηση και πολιτικά και οικονομικά στο κοσυφοπαίδιο Γι' αυτό έχω υπερψηφίσει αυτή την έκθεση. Μάμικινς. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε η Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κωσυφοπεδίου αν ε, θα οδηγήσει ε, σε μια περαιτέρω σταθεροποίηση τη περιοχή των Βαλκανίων και αυτό συνιστά μείζωνα επένδυση ε, στον δρόμο της ένταξης του Κωσυφοπεδίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελπίζω όμω να τονώσει και την ανάπτυξη στη χώρα αλλά και να βελτιώσει τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα. Πέραν όλων αυτών. Θέλω να πω ότι η σημερινή ψηφοφορία είναι πάρα πολύ σημαντική και για έναν ακόμη λόγο. Για να ληφθεί υπόψη και η κατάσταση της σερβικής μειονότητας στο βόρειο τμήμα της χώρας. Η ε, συμφωνία όμως ε, δεν ξέρουμε κατά πόσο θα μπορέσει να προωθήσει ε, κάτι τέτοιο. Επειδή όμω θεωρώ ότι θα μπορούσε να οδηγήσει στη συμβουλή μεταξύ και αρμονική συμβουλή μεταξύ των διαφόρων, την ψήφισα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπω είπε και είπατε εκπρόσωπο κυρία Μαγκερίνη για τη συμφωνία αυτή τη Ευρωπαϊκή Ένωση του Κωσυφοπεδίου, ξεκινάει έτσι μια νέα φάση στι σχέσει μεταξύ 28 κρατών μελών και τη χώρα αυτή. Η συμφωνία είναι μια σημαντική συμβολή στη σταθεροποίηση και την ευημερία στην όλη περιοχή, προσφέροντα κίνητρα για να γίνουν οι απαραίτητε μεταρρυθμίσει και να υπάρξει βιώσιμη και σταθερή ανάπτυξη. Χρειάζονται αυτέ οι μεταρρυθμίσει για να δημιουργηθούν εμπορικέ ευκαιρίε επενδύσεων. Η κυβέρνηση του Κοσφοπεδίου συνεχίζει την προσπάθεια των μεταρρυθμίσεων και την προσπάθεια να εξυγχρονιστεί και να αναπτυχθεί από άποψη οικονομική και εμπορική για να προσφέρει ένα καλύτερο μέλλον στου πολίτε τη. Το Κοσφοπέδιο πρέπει να αντιμετωπίσει ακόμη πολλά προβλήματα. Ελπίζω λοιπόν η κυβέρνηση να κάνει τι σωστέ και τολμηρέ επιλογέ που χρειάζονται για να προχωρήσουμε επιτυχία στι διαπραγματεύσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε κύριε Καπούτο. Ο κύριο Πόσπισιλ. Για ένα λεπτό κι εσεί. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και εγώ υπερψήφισα την ε, προτινόμενη συμφωνία με το κόμμα το γεγονό ότι υπάρχουν πολλέ χώρε στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν έχουν αναγνωρίσει το κοσμοπέδιο ω ανεξάρτητο κράτο. Είναι ενδιαφέρον αυτό που είπαν οι προλαλήσαντε, ότι έχει σταθεροποιηθεί η κατάσταση εκεί και αυτό βολτιώνει τη δυνατότητα των χωρών τη γειτονιά του του κοσμοπέδιου να έχουν μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη και καλύτερη προοπτική να γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο μέλλον ο δρόμος του κοσυφοπεδίου στην προς την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα είναι σύντομος, δεν θα είναι απλός. Θα χρειαστεί πολλής χρόνος για να γίνουν οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις στο κοσυφοπέδιο για την κρατική μηχανή και το σύνολο τη κοινωνία. Αυτό είναι προφανέ, αλλά σήμερα θέλουμε να στείλουμε σαφέ μήνυμα προ το Κωσυφοπέδιο τονίζοντα ότι πρέπει να υπάρξει καλύτερη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει μακροχρόνια να εξασφαλίσουν την ένταξή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα Βαλκάνια και το σύνολο τη Ευρώπη. Αυτό είναι πάρα πολύ και αυτό υπερψήφισε. Ευχαριστώ. Σόγκορ. Ένα λεπτό επίσης. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης με το Κοσφοπέδιο ε, θα τεθεί τώρα σε εφαρμογή αυτό είναι κάτι το οποίο μου δίνει την ευκαιρία να παροτρύνω τα πέντε κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχουν αναγνωρίσει επίσημα στο Κωσυφοπέδιο, μεταξύ των οποίων και η δική μου χώρα η Ρουμανία, να το πράξουν. συγχρόνως η ενσωμάτωση και η ολοκλήρωση των υπολείπων χωρών των Δυτικών Βαλκανίων αυτή τη στιγμή είναι αδύνατο να λάβει χώρα χωρίς να λυθεί το πρόβλημα της συνδύωσης των διαφόρων εθνοτικών ομάδων. Πρέπει να το προωθήσουμε αυτό. Δεν το λέει αυτό τώρα η συμφωνία. Έχουν κάποιες, έχει κάποιες γενικές μνήες. Η εμπειρία δείχνει όμως ότι αυτά τα οποία λέει δεν επαρκούν στα κράτη-μέλη μας. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κάτι το οποίο δεν γίνεται πάντα, γιατί τα κράτη-μέλη δεν κάνουν πάντα τους απαραίτητους τι απαραίτητε ενέργειε και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δίνει σημασία παρά το γεγονό ότι αυτό αφορά 40 εκατομμύρια πολιτών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι εύκολο να είναι κανεί μέλο μια μειονότητα στο κοσφουπέδιο. Θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Πόλτσακ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η αυτοδιάθεση όλων των εθνών είναι ένα από τα πολλά σημαντικά στοιχεία που συμπεριλαμβάνονται στη χάρτα του ΟΗΕ για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Για παράδειγμα, το πρόβλημα είναι ότι ορισμένες χώρες δυσκολεύονται διότι δεν αναγνωρίζουν τα δικαιώματα άλλων εθνών. Εγώ πρέπει να πω ότι το κοσυφοπέδιο έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός εθνικού κράτους. Ακόμη και αναγυρώνται κάποια ζητήματα, αυτό δεν το αρνούμε, αλλά δεν θα ήθελα να ε, προσπαθήσω να αντικρούσω τα επιχειρήματα της κυρίας Μορβάη. Και το κοσμοπέδιο έχει τις ιδιαιτερότητές του και αυτό ισχύει για όλες τις χώρες της Επίρου μας. Γι' αυτό θα ε, συμφωνήσω πολύ με τον κύριο Σόγκορ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κλείνουμε τις απεξηγήσεις ψήφου για τις ελεύθερες συναλλαγές με την, ε, για την έκθεση αυτή. Και περνάμε στην ε, Γεωργία, Μολδαβία και Ουκρανία και τι Φερικέ Ξεπατού Συμφωνίε Ελευθερών Συναλλαγών με αυτέ. Η κυρία Ντάνοκα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ καταψήφισα αυτό το ψήφισμα συζητώντα ε, για το θέμα σήμερα. Ε, ακούσαμε πράγματα που μπορεί να δείχνουν και ότι υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά, κάποια ψεύδια ακούστηκαν. Ε, στην παράγραφο 34 που εγκρίθηκε σήμερα για τον Ντομπάς και για μια άλλη περιοχή ε, για το Λουγκάνς και τον Ντονέσκα. Λέτε ότι είναι κατεχόμενα, μα από ποιους. Τοπικοί πληθυσμοί κατέχουν εντό αγωγικών στον Ντανιέσκ. Κινδυνεύουν οι πολίτες Ποιοι είναι αυτοί που ε, κατέχουν μία 17χρονη η οποία ε, έχασε ε, τα δύο πόδια και χέρια της μετά από φοβιστική απόδειξη που σε ένα λεωφορείο. Και σίγουρα είναι σημαντικό το ότι βοηθήσαμε να αποκτήσει τεχνητά μέλη η συγκεκριμένη κοπέλα Γιούλια, αλλά υπάρχουν και χιλιάδες άλλοι στη θέση αυτή. Ευχαριστούμε ο κύριος Γιάρια ένα λεπτό. Ε, ε, ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Προέρχομαι από την Ουγγαρία και είμαι μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εκπροσωπώ την Ουγγαρία όπως ξέρετε. Όταν πρέπει να ψηφίσω για συμφωνία σύνδεσης και σταθεροποίησης εγώ σκέφτομαι περισσότερο για τα ανθρώπινα δικαιώματα των Ούγγρων που ζουν στην Ουγγαρία. Οι Ούγγροι οι Ούγγροι της, περιοχής, της υποκαρπάθειας περιοχής δεν μπορούν να μιλήσουν για αυτονομία ή για αυτοδιάθεση. Αυτό είναι σε αντίθεση με αυτά που είδαμε όταν μιλήσαμε για το Κωσυφοπέδιο προηγουμένως. Σε κάθε σημαντικό έγγραφο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λέγεται ότι η αυτοδιάθεση είναι συλλογικό ανθρώπινο δικαίωμα. Αυτό είναι πολύ βασικό. Αν το πείτε όμως αυτό εντορία φωνή στην ε, Ουκρανία και αναφερθείτε στα δικαιώματα των Ούγγρων για αυτονομία, τότε αυτό θα οδηγήσει σε διώξεις και πάρα πολύ άμεσες αντιδράσεις και κολασμό. Ένα μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, παραδείγματος χάρη, εξεδιώχθη από την Ουκρανία για αυτό το λόγο. Δεν υπάρχει σεβασμός λοιπόν για τα δικαιώματα των μειονοτήτων και για την αυτονομία και αυτοδιάσκη γι' αυτό κατεψήφισα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριο Γιάρ. Ο κύριο Γιάρ. Μπορεί κανεί να βρει λόγου για να καταψηφίσει αυτή την έκθεση, προφανώ. Το κατανοώ αλλά βρισκόμαστε μέσα στα πλαίσια μια διαδικασία που νομίζω πρέπει να την αντιμετωπίσουμε με αισιοδοξία. Νομίζω ότι η οικονομική συνεργασία πολλέ φορέ αποφέρει καλύτερου καρπού από την πολιτική, δημιουργεί αυτή η συμφωνία επαφέ και μπορεί να βελτιώσει την πολιτικο-οικονομική εξέλιξη στο μέλλον. Όλα αυτά είναι η δημιουργία εμπιστοσύνης και ελπίδος στις χώρες αυτές. Και όπως είπα και προηγουμένως στη συζήτηση για το κοσφοπέδιο, αυτό από μόνο του είναι επαρκές για να εξασφαλίσει μια θετική ψήφο και να θέλω να εκφράσω την ε, ελπίδα μου για μια πιο θετική διαδικασία. Ο αποκλεισμό είναι κάτι το οποίο είναι το αντίθετο από αυτά που θέλουμε. Παρ' όλα αυτά φυσικά θέλουμε να παρακολουθήσουμε προσεκτικά την ε, διαδικασία αυτή και να δούμε τι θα προκύψει στο τέλος και είμαι μαζί με όλους αυτούς που θέλουν τη δημοκρατικοποίηση. Μανίκινς για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Όταν ο εισηγητής ε, για τη γεωργία ε, γίνονταν όλα αυτά τότε και τα είχα παρακολουθήσει εκ του σύνεγγυς και το τι σημαίνει στην ευρύτερη περιοχή. Γι' αυτό πρέπει να σας πω ότι χαίρομαι πολύ που βλέπω ότι υπάρχουν ε, πολλές ενέργειες που θα μπορούσαν να φέρουν πιο κοντά τη Γεωργία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία, πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι' αυτό θεωρώ ότι είναι αξιέπαινο ε, να συναυθεί Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών και να μπορούν και οι Ουκρανοί χωρίς βίζα να μπορούν να ταξιδεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρόλα αυτά αυτά Καταψήφισα την έκθεση και γιατί το έκανα αυτό. Γιατί ήθελα να καταλάβω γιατί χρησιμοποιούμε αυτή τη γλώσσα σε βάρος της Ρωσίας. Πραγματικά πιστεύουμε ότι θα έρθει να στήσει γνώμη μετά από αυτό το ψήφισμα η Ρωσία. Πρέπει να έχουμε ένα επικοδομητικό διάλογο με τη χώρα αυτή και δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε τέτοια φρασιολογία στο ψήφισμά μας. Ευχαριστώ ο κύριος Καπούτο. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Συμφωνία Σύνδεση Ελεύθερων Συναλλαγών μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση, Γεωργία, Μολδαβία και Ουκρανία είναι αναγνώριση τη αξιοσημείωτη πρόοδου που έχουν καταβάλει οι χώρε αυτέ προκειμένου να καταλήξουν σε ένα φυσικό και λογικό αποτέλεσμα τη πορεία που έχουν ξεκινήσει πριν από μια δεκαετία. Οι συμφωνίε αυτέ είναι προ συμφέρον όλων και είναι ένα σημείο αναφορά για την πολιτική μα γειτονία προ τα ανατολικά. Θα πρέπει να συνεχίσουμε στον δρόμο των μεταρρυθμίσεων ε, και να, προωθήσουμε, να παροτρύνουμε τις χώρες αυτές να ακολουθούσαν αυτή την οδό για την οικονομική και κοινωνική του ανάπτυξη. Θα πρέπει την ιστορική πολιτική και τον εξυγχρονισμό των χωρών αυτών να τι ευνοήσουμε, προκειμένου να αναπτυχθούν χωρί πρόβλημα οι εταίροι μα και να υπάρχει εθνική συνένεση για τα απαραίτητα μέτρα ώστε να υπάρξει βιώσιμη ε, και ουσιαστική αλλαγή. Η Συμφωνία Σύνδεσης μπορεί να φέρει τις απαραίτητες πολιτικές αλλαγές και την ανάληψη πρωτοβουλειών στο εσωτερικό των χρόνων αυτών. Η διαδικασία μεταρρυθμίσεως μπορεί να οδηγήσει στην ταμπή ε, ε, στις χώρες αυτές με τη διοικητική δικαστικό του σύστημα και το δικαστικό σύστημα να ε, μεταρρυθμίζονται. Ευχαριστούμε κύριο Πόσπιση. Ευχαριστώ Πρόεδρε ε, στη Δημοκρατία της Τσεχίας, την οποία εκπροσωπώ. Έχουμε τραγικές εμπειρίες από το κομμουνιστικό καθεστώς. Γι' αυτό πάντοτε θα υποστηρίζω τα σχέδια γειτονία προ Ανατολά και οποιαδήποτε μορφή οικονομική συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τι πρώην χώρε τη Έσου Εδώ οι λόγοι είναι γεωπολιτικοί. Η Ρωσία ουδέποτε κοιμάται. Και με, υπό αυτήν την έννοια έχει λόγους να επιδιώκει τα συμφέροντά της στις πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες. Καθημερινά βλέπουμε τι προβλήματα αντιμετωπίζει η Μολδαβία, λόγου χάρη. Πρέπει τις πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες, να τις υποστηρίξουμε, να τις ε, αντιλαμβανόμαστε ως εταίρους και να συνεργαζόμαστε μαζί τους. Πρέπει να βελτιώσουμε και την οικονομική τους κατάσταση, αλλά όπως προείπα, ο λόγος που στηρίζω αυτές τις συμφωνίες είναι γεωπολιτικός. Το να είναι εταίρος για πρώην ε, Σοβιετική Δημοκρατία σε άλλες συμφωνίες που δεν εμπλέκεται η Ρωσία είναι πολύ σημαντικό. Ευχαριστούμε Σόιντροβα. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, εγώ ήμουν υπέρ του ψηφίσματος ε, για τις φωνές ε, σύνδεσης ε, με Γεωργία, Μολδαβία και Ουκρανία. Δεν στήριζα τις προτάσεις κομμουνιστικών κομμάτων που υπονομεύουν δημοκρατικά εκλεγμένες κυβερνήσεις και συγκεκριμένα υποσκάπτουν ε, την προσχώρηση, την, μάλλον το, την προσέγγιση της Μολδαβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντως, ε, ε, αν και σπάνια συμβαίνει, ικανοποιήθηκα τις προτάσεις του Επιτρόπου Χαν και της Κομισιόν σε ό,τι αφορά τις θεωρήσεις για τους υπηκόους της Ουκρανίας. Και είναι και κάτι που ικανοποιεί και τη χώρα, η οποία έχει υψηλές προσδοκίες από την απελευθέρωση του συστήματος θεωρήσεων και τους δίνει νέα όθηση και νέο ενθουσιασμό. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω τον Επιτρόπο και την Κομισιόν γενικά. Άνεμανς. Θα ήθελα να κάνω σαφές γιατί εγώ καταψήφισα αυτή τη συμφωνία σύνδεσης με την Ουκρανία. Δεν εμπλέκεται το θέμα της, ε, των ελευθέρων συναλλαγών, αλλά τη γεωπολιτική δύναμη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παίζει ένα δύσκολο και επικίνδυνο παιχνίδι όταν παρεμβαίνει σε αυτή την περιοχή και δημιουργεί αντιπαραθέσει. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να έχει ελεύθερο εμπόριο, πρέπει να σταματήσει το εμπάργκο κατά τη Ρωσία που είχε τόσο αρνητικά αποτελέσματα στου Ευρωπαίου γεωργού. Δεν πρέπει να οξύνουμε περισσότερο τα προβλήματα με, στην περίπτωση αυτή με την Ουκρανία. Θέλουμε να υποστηρίξουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά το να προετοιμάσουμε την ε, Ουκρανία ε, για να έρθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα δημιουργήσει ένα νέο ψυχρό πόλεμο. Πόλτσακ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Εγώ υπεστήριζα την συμφωνία αυτή σύνδεσης και αυτά είναι σημαντικά οικονομικά θέματα που αντιμετωπίσουμε για αυτές τις συμφωνίες. Δεν θέλω να διαμφισβητήσω τα δικαιώματα των εθνικών μειονοτήτων, αλλά εδώ εμπλέκονται πολύ περισσότερα θέματα. Για να μπορέσουμε εμείς τώρα να καθορίσουμε το πώς μια άλλη χώρα θα πρέπει να οργανωθεί σε ό,τι αφορά τα εσωτερικά της θέματα δημοκρατικά δικαιώματα μειονοτήτων και αυτονομία, αυτό δεν νομίζω ότι είναι δικό μας θέμα. Για την Μολδαβία, <clears throat> εδώ έχω κάποιες ε, αμφιβολίες και συνεχίζω αυτά που είπε ο κύριος Πεσπέλ. Ένα ερώτημα πρέπει να ρωτήσουμε τους εαυτούς μας είναι το εξής. Κινδυνεύουμε να είμαστε ε, μάρτυρες μιας κατάστασης όπου οι Ρώσοι ολιγάρχες θα ελέγξουν τις, τους κυβερνητικούς συνασπισμούς ακόμα και την αντιπολίτευση στις χώρες αυτές. Αυτό πρέπει να το παρακολουθήσουμε από πολύ κοντά. Ευχαριστώ. Περνάμε στις επεξηγήσεις ψήφων για τη ρήτρα αμοιβαίας άμυνας. Η κυρία Μορβάη για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η ρήτρα μηδέας άμυνας που αφορά το θέμα αυτό είναι ένα σημείο για το οποίο υποβλήθηκαν πολλά ενδιαφέροντα ψηφά από την ομάδα EFTD όπου αναφέρεται στο κείμενό μας ότι ε, οι πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις στην κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αυτό αναφέρεται στο σημείο ε, ε, επιβάλλουν την ανταλλαγή μυστικών πληροφοριών και τη συνεργασία μεταξύ των μυστικών υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί αποδείχθηκε ως τώρα ανεπαρκής. Υπήρξαν σοβαρές ελλείψεις και κενά στον τομέα αυτό, το οποίο το αναφέρει και το ψήφισμα των Πρασίνων, Μιλάει για το εμπόριο όπλων. Επιτέλους αρχίσαμε να μιλάμε για την ουσία και όχι να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας ή να υπεκφεύγουμε. Οι μυστικές υπηρεσίες δεν έχουν τίποτε ε, να κάνουν ε, με, την τρομοκρατία και δεν είναι αυτό απάντηση στη δημοκρατική απειλή. Ο κύριος Γιούρεκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι η ρήτρα αμοιβαίας άμυνας θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στην έκφραση της αλληλεγγύης στο ΝΑΤΟ, διότι τρία τέταρτα των κρατών μελών είναι και μέλη του ΝΑΤΟ. Θα πρέπει επίσης να αντικατοπτρίζεται στην κινητοποίησή μας όσον αφορά την πρώτη προτεραιότητά μας, την ασφάλεια. Νομίζω ότι εάν 75% των κρατών μελών συμμετέχουν έτσι και αλλιώ στο ΝΑΤΟ, ε, νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο να εξασφαλίσουμε περισσότερη ασφάλεια και για την Λετωνία και την Εστονία. Εάν μιλάμε για αμοιβαία άμυνα και ασφάλεια, θα πρέπει να είμαστε πιο δραστηροί σε επίπεδο ΝΑΤΟ και να απόσχουμε από τον πολλαπλασιασμό δηλώσεων επί χάρτου ή όλη αυτή τη σχιζοφρένεια που μας έχει ε, καταβάλει στην ε, Ευρωπα... μας έχει κυριεύσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προτού γίνουμε κάτι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπήρξαμε μέλη μιας συμμαχίας που θα μπορούσε να αναλάβει δράση όταν έπρεπε να εξασφαλίσει την προστασία μας. Ευχαριστούμε, μα σε ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μετά από τα τρομερά γεγονότα του Παρισιού της τρομοκρατικές επιθέσεις του Νοεμβρίου, η Γαλλία έγινε η πρώτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ήθελε να υπάρξει η εφαρμογή του άρθρου 42.7 και όχι του άρθρου 2.27 της ρήτας αλληλεγγύης. Τα περισσότερα κράτη-μέλη έχουν ανταποκριθεί στο αίτημα της Γαλλίας. Αυτό είναι φυσιολογικό, γιατί είναι αδύνατο να αντιμετωπιστεί η τρομοκρατία μόνο σε μία χώρα. Πρέπει να καταδείξουμε την αλληλεγγύη μας σε όλες τις πτυχές και εκφάνσεις της και φαίνεται ότι θα πρέπει να αποδώσουμε την πρέπουσα σημασία στον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσει η ενεργοποίηση του αρθρού 42 εάν αυτό καταστεί απαραίτητο. Γιατί κάτι αντίστοιχο, ελπίζω όχι, μπορεί να συμβεί σε άλλες χώρες. Ο μηχανισμός αυτός πρέπει να είναι σωστός από νομική άποψη. Ευχαριστώ Καπούτο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η αλληλεγγύη, η βοήθεια και η αλληλοβοήθεια των κρατών μελών θα πρέπει να εξασφαλίζουν την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάντως καλωσορίζουμε την ομόφωνη στήριξη της Γαλλίας από τα υπόλοιπα κράτη-μέλη και την προθυμία τους να προσφέρουν την απαραίτητη βοήθεια μετά την ε, επίκληση τη ε, ρήτρα αμοιβαία άμυνα από την ίδια τη Γαλλία μετά τι επιθέσει στο Παρίσι. Πάντω, αυτή τη στιγμή λείπουν οι πρακτικέ διαδικασίε για να έχουμε μια πρακτική ενεργοποίηση, μια γρήγορη ενεργοποίηση, οπότε να κάτω το επικαλεστεί τη ρήτρα αμοιβαία άμυνα. Η είπατε εκπρόσωπος ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κυρία Μογκερίνη, εργάζεται αδιάκοπα για να βελτιώσει την ε, ταχύτερη ενεργοποίηση της ρήτρα αυτής στο μέλλον. Θα πρέπει να λάβουμε τέτοιες αποφάσεις μαζί με το Συμβούλιο για να μπορούμε να προστατεύσουμε το κάτω μέλος που δέχεται επίθεση. Θα πρέπει η ρήτρα αυτή να επιτρέπει σε όλο, σε οποιονδήποτε την επικαλεστεί, να αξιοποιεί στην ε, να αξιοποιεί την πλήρη, τις πλήρες δυνατότητες που προσφέρει η ρήτρα αυτή. Και... Λοιπόν, ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ υπερψήφισα το ψήφισμα αυτό, διότι και εγώ πιστεύω ότι είμαστε σε πόλεμο κατά της τρομοκρατίας όλοι και όχι μόνο η Γαλλία που δέχτηκε τις επιθέσεις τον προηγούμενο Νοέμβριο. Όχι. Ο ευρωπαϊκός πολιτισμός στο σύνολό του είναι αντιμέτωπος με την τρομοκρατία. Το ίδιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήδη οι συνάδελφοι ανέφεραν ότι από την ε, μία ε, πρώτη φορά χρησιμοποιείται αυτό το μέσο ε, δυνάμει του άρθρου 42 της συνθήκης της Λισαβόνας. Πρέπει να δούμε λοιπόν πώς θα κινηθούμε και πώς θα εφαρμόσουμε πρακτικά το ψήφισμα και να μην μείνουμε ε, στα μεγάλα λόγια όπου θα δεκηρύσουμε την αλληλεγγύη και την αμοιβαία άμυνα και θα μείνουμε εκεί. Η τσεχική δημοκρατία προσπαθεί να βοηθήσει πραγματικά τη Γαλλία. Γι' αυτό συνεργαζόμαστε και σε πολλές τους ε, ε, δράσεις εκεί στο Μαλί. Αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε ένα ειδικό χώρο για αυτό το μηχανισμό. Το 79, ξέρετε κύριε Πρόεδρε, λέει ο κύριος Γόλφ, υπερψήφισαν την ε, Ένωση ως έναν ε, οργανισμό ελεύθερου εμπορίου και τώρα θα ψηφίσουμε με δημοσίευμα θέλουμε να παραμείνουμε σε αυτόν τον οργανισμό, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τώρα μας ζητείτε να έχουμε ουσιαστικά ένα ευρωπαϊκό ε, στρατό, αυτή την αμοιβαία άμυνα εμείς που δεν θέλαμε να μπούμε σε αυτή την εμπορική ένωση, δεν θέλουμε να μπούμε σε μια αυτοκρατορία που θα θέλει μόνο και μόνο να επεκτείνει τα σύνορά της ε, και ε, δεν θέλουμε να ε, δίνουμε ένα ράπισμα στη ΣΥΠΑ και στο ΝΑΤΟ που έχουν κρατήσει ζωντανή την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί με αυτό θέλουμε να δημιουργήσουμε τελικά μια Ευρωπαϊκή Συμμαχία και ένα Ευρωπαϊκό στρατό. Δεν είμαι υπέρ η Ευρωπαϊκή Ένωση να την επιλογή να γίνει αυτοκρατορία και να έχει το δικό της στρατό. Εγώ πιστεύω στην ελευθερία και τη δημοκρατία και στα κράτη-έθνη και πιστεύω ότι οι Βρετανοί θα ψηφίσουν ε, η χώρα τους να φύγει από την Ένωση γιατί αυτό που επιθυμώ εγώ το επιθυμούν και οι ίδιοι. Ευχαριστώ. Ωραία, και τώρα συνεχίζουμε με την ημερήσια διάταξη. Επεξηγήσει ψήφου για τι προτεραιότητε τη Ευρωπαϊκή Ένωση ενώπιση των συνόδων του UNHCRC για το 2016. Το λόγο έχει ζητήσει η κυρία Μορβάη, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει κυρία Μορβάη. Όταν πρόκειται για τις προτεραιότητες για την υπάτη αρμοστία των Ηνωμένων Εθνών, εγώ δεν μπόρεσα να υπερψηφίσω αυτή την έκθεση, γιατί κάθε ψήφισμα τονίζει ότι πόσο σημαντικό είναι να εξασφαλίσουμε τα δικαιώματα των πολιτών και τα οικονομικά τους δικαιώματα και τα κοινωνικά τους δικαιώματα και να πούμε ότι αυτά είναι αναπαλωτρίωτα. Τώρα όμως που είμαι μέλος του Κοινοβουλίου εδώ και 6,5 χρόνια και έχω δει τι γίνεται στη δική μου χώρα και τι γίνεται και στην Πολωνία που και οι δύο χώρες έχουν κατασυκοφαντηθεί για υποτιθέμενες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν μπορεί κανείς να ρωτήσει πώς είναι δυνατόν ένας πυροσβέστης ή ένας δάσκαλος στην Ουγγαρία να παίρνει μόνο 20% των αποδοχών ενός αντίστοιχου εργαζόμενου στην ε, Δυτική Ευρώπη. Όταν λοιπόν αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα μπορούμε να συζητήσουμε τα υπόλοιπα. Ευχαριστώ ένα λεπτό κύριε Μπολόπες Μπερμέχου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το αίτημα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς που ψηφίσαμε εμείς ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση να υποστηρίξει τη θέση η οποία έχει εγκριθεί στο παρελθόν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δηλαδή ότι θα πρέπει να υπάρξει έρευνα για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Δυτική Σαχάρα. Ότι το βασίλειο του Μαρόκου θα πρέπει να απελευθερώσει τους πολιτικούς κρατούμενους των Σαχαραούι. Να επιτρέψει την ελεύθερη πρόσβαση στη, στα κατεχόμενα εδάφη της Δυτικής Σαχάρας. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να εθελοτυφλούμε σε μια κατάσταση η οποία μέρα με τη μέρα οξύνεται και επιδεινώνεται. Και το Μαρόκο κάνει ό,τι μπορεί για να κουκουλώσει. Όπως φάνηκε με την πρόσφατη ε, εκδίωξη πολλών ε, παρατηρητών ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την Ορβηγία και τη Σουηδία. Ζητούμε και πάλι να απελευθερωθούν οι πολιτικοί <clears throat> κρατούμενοι από τη Δυτική Σαχάρα και ζητούμε από την Ισπανία να δώσει στον Χασάν και στους συντρόφους τους το πολιτικό άσυλο. Ζητούμε να τονίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την αλληλεγγύη του με τους άνεργους Σαχαραούι που ασκούν ε, απεργία πείνας και να υποστηρίξουμε αυτούς που αγωνίστηκαν εναντίον της κατοχής. Γιούρεκ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τα τελευταία δύο χρόνια οι Σλοβάκοι, οι Σλοβαίνοι και οι Κροάτες οργάνωσαν δημοψηφίσματα με θέμα την σύνθεση της οικογένειας κατά φύση και μετά από τα αιτήματα των κινημάτων των ομοφιλοφίλων παρόμοιους κανόνες βρίσκουμε στα συντάγματα της Λιθουανίας και της Ουγγαρίας όμως και πάλι το Κοινοβούλιο σήμερα ψήφισε υπέρ της αποδοχής τέτοιων ετοιμάτων. Αντί στον ΟΗΕ να παρουσιάσει τις θέσεις όλων των χωρών, ή τουλάχιστον να σεβαστεί τις απόψεις των χωρών αυτών, όπως εκφράστηκαν σε εθνικά δημοψηφίσματα, το Ευρωκοινοβούλιο θέλει Ευρωπαϊκή Ένωση να μας αλλάξει, όχι να μας εκπροσωπεί, να μας αλλοιώσει. Εδώ η μέγιστη απειλή για τη δημοκρατία μας είναι οι ίδιε οι πολιτικέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε Μαμίκινς για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Οι εθνικές και θρησκευτικέ μειονότητε και παραβράστων των δικαιωμάτων τους αλλά έχουμε και άλλους, ε, τα παιδιά, τις γυναίκες, ε, και όλα αυτά δείχνουν ότι είναι πολύ σημαντικό και εμείς να είμαστε πολύ δραστήριοι στο πλαίσιο των συνεδριάσεων του Συμβουλίου τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του ΟΗΕ. Πολλά πρέπει να λάβουμε υπόψη και πολλές τις μέσεις πρέπει να τηρηθούν. Πάντως, Υπάρχει πρόβλημα ε, στο Συμβούλιο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων να ε, μπλοκάρουν ε, τις ψηφοφορίες. Υπάρχουν κάποιες χώρες που έχουν κάνει μια συμμαχία, παραδείγματο χάρη στηρίζεται το Ισραήλ, η Σαουδική Αραβία μπορεί να προεδρεύσει επίσης μιας δέσμης χωρών που θα ήταν κατά του Ισραήλ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σόντροβα. Τέψατε με συντομία. Να σα εξηγήσω γιατί δεν ψήφισα υπέρ τη γνωμοδότηση αυτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τι προτεραιότητε τη Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο των συνεδριάσεων του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το 2016. Αυτό το ψήφισμα περιλαμβάνει ρήτρε με τι οποίε δεν μπορώ να συμφωνήσω, ε, δεν μου το επιτρέπει η συνείδησή μου. Υπάρχει μια ακροφιλελεύθερη ε, αντίληψη ε, σε ό,τι αφορά τα γενετικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα που ουσιαστικά κάνει την ε, έκτρωση τη μόνη λύση σε οποιοδήποτε προγενετικό πρόβλημα εντοπιστεί. Βέβαια η άποψή μου αυτή είναι μειονοτική ή όταν μίλησα για τους Ισραηλινούς επικισμούς ως κάτι που υπονομεύει την ειρηνευτική ε, διαδικασία. Ε, πάλι κάποιοι ψευδείς ισχυρισμοί περιλαμβάνονται στο ψήφισμα, εξού και χρειάστηκε να το καταψηφίσω. Ευχαριστώ. Και τώρα επεξηγήσει ψήφου για τι δραστηριότητε τη Επιτροπή Αναφορών 2014. Η κυρία Μορβάη έχει ζητήσει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η έκθεση αυτή για το έργο της Επιτροπής Αναφορών προκάλεσε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση εδώ. Και είπα κατά τη διάρκεια της συζήτησης ότι ένα πολύ απλοϊκό ε, κείμενο μεσής σελίδας ετοιμάστηκε για να απαντήσει στις 15 σελίδες Ούγκρων αναφερόντων ε, τα τελευταία χρόνια. Ε, νομίζω ότι την 15 σέλιδη αναφορά τους οι Ούγγροι πολίτες δεν την έδωσαν, δεν την έδωσαν στον κλητήρα της αίθουσα. ακόμη και εκείνο θα έχει ετοιμάσει μια πιο, ε, πιο λεπτομερή απάντηση από ό,τι έκανε η Επιτροπή Αναφορών. Αυτό είναι πραγματικά το παράδοξο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μένα και είναι και μαύρο το χιούμορ ε, όσων λένε ότι εργάζονται εδώ Εργάζονται για να βελτιώσουν τη ζωή των πολιτών μας. Εάν αυτό θεωρούν δουλειά και έτσι αντιμετωπίζουν τις ανασφορές, τις αναφορές, έτσι θα καταντήσουν και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θεσμικά της όργανα. Ε, ε, έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα. Κανείς δεν έχει ρωτήσει τους ανθρώπους μονομένα αν θέλουν να είναι μέλη τη Ένωσης και τη Επιτροπής Αναφορών. Ευχαριστούμε. Δεν είναι εδώ ο κ. Ντάλι, οπότε ο Μπενίτο Λουάγκα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Οι υποδέμος πάντα έχουν υποστηρίξει τη συμμετοχή των πολιτών και επομένως δίνουμε μεγάλη, δυνα... Ε, μεγάλη υποστηρίξη στο δικαίωμα της αναφοράς αλλά επίση μας ενδιαφέρει και η συμμετοχή των πολιτών στην πολιτική συζήτηση. Δύο γεγονότα. Πρώτα, η Ισπανία είναι η χώρα από την οποία έχουμε τις περισσότερες αναφορές. Αυτό καταδεικνύει το γεγονός ότι υπάρχει μια πραγματική κοινωνική κίνηση στην Ισπανία. Δεύτερον, ότι κυρίως αφορούν θέματα ενέργειας και περιβάλλοντος, δηλαδή για την υδροενεργομάτωση και τις έρευνες για πετρέλαιο στα Κανάρια. Εμείς τονίζουμε ότι η ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική αυτή τη στιγμή παραμένει αντιδημοκρατική. Μονάχα τρεις από τις 31 Πρωτοβουλίε πολιτών έχουν καταλήξει και προ το παρόν μόνο μία από αυτέ έχει φτάσει στο σημείο που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αρχίσει να κάνει κάτι για αυτήν. Φαίνεται από όλε τι πλευρές τη Ευρώπη ότι υπάρχει μια διεκδίκηση μια πραγματικά δημοκρατική και συμμετοχικής Ευρώπη. Και αυτό είναι εφικτό αγαπητοί συνάδελφοι. Ευχαριστώ κύριο Γιάρη για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δύο πράγματα θέλω να πω ως συντονιστής για το ΕΛΚ της Επιτροπής Αναφορών. Πρώτα απ' όλα εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα για την μεγάλη υποστήριξη που έλαβε η έκθεση της κυρία Φέντουγκερ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό είναι ένα καλό μήνυμα για τη συνέχιση τη εργασία μας. Δεύτερον όμω πρέπει να αναφέρω πράγματα τα οποία δεν με έχουν ικανοποιήσει και εγώ έχω αγωνιστεί προσωπικά για το να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια στην Επιτροπή ε, αναφορών γνωρίζω την ε, σημασία της γραμματείας αυτής της Επιτροπής, αλλά το θέμα της ε, εμπειρογνωμοσύνη τους θα απαιτούσε και περισσότερο προσωπικό. Δεν είναι λοιπόν ούτε λυσιτελές ούτε δίκαιο αυτό που γίνεται στην, Ευρωπαϊκή, στην Επιτροπή Αναφορών. Είναι απαραίτητο να εξασφαλίσουμε τις προϋποθέσεις για να γίνεται μια συζήτηση επί της ουσίας Παρά το γεγονό βέβαια ότι αυτά δεν με ικανοποιούν, εγώ ε, υπερψηφίζω αυτή την έκθεση. Μα μη Ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Η Επιτροπή Αναφορών έχει ένα όνομα. Και είναι πολύ σημαντικό που μπορούν οι πολίτες να απευθύνονται το 2014 ήταν μικρότερες οι αναφορές, λιγότερες από το προηγούμενο έτος, αλλά ε, η γενική τάση είναι αυξητική και αυτό είναι καλό γιατί σημαίνει ότι είναι καλύτερα ενημερωμένοι πολίτες σε σχέση με τις δράσεις της Ένωσης. Όμως πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι περίπου το 40% των αναφορών κρίνονται μη παραδεκτές. Άρα δεν υπάρχει τελικά επαρκής ενημέρωση δεν γνωρίζουν δηλαδή ε, οι συντάκτες γιατί πρέπει να ε, συντάξουν αναφορές, γιατί αντικείμενο κάθε φορά. Άρα πρέπει να βελτιώσουμε τις ενημερωτικές εκστρατείες, ε, να αυξήσουμε την πληροφόρηση, να διαδώσουμε την πληροφόρηση και να ζητήσουμε από τους πολίτες να καταθέτουν συχνά αναφορές. Ευχαριστούμε κύριε Μαμίκιν. Ήταν η τελευταία παρέμβαση για σήμερα το πρωί. Ε, διακόπτεται η σύνοδος μέχρι τις 3.